Uh, Χθες ξέχασα να υπογράψω. Αυτό είναι. Απλά. Ήμουν εδώ. Ξέχασα να υπογράψω. Έχω, έχω υπογράψει ήδη στον κατάλογο παρουσιών της συνεδρίας μας. Μην νομίζετε ότι με τεμπέλης. Απλά ξέχασα να υπογράψω. Να γραφεί παρακαλώ στα πρακτικά. Ωραία. Θα το σημειώσουμε κύριε Σλίτελη Πρόεδρος. Η κυρία Ντεκεζέρ έχει δει στο λόγο. Προσπαθώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω, επειδή δεν είναι πήγον σε αυτή την Σύνοδο Λομέλειας, να παρέμβουμε ώστε να στραφεί ο πρόεδρος Σούλτς προς τις αρχές και να απευθύνει έκκληση να μην εκτελεστεί ο κύριος Μπαλουάν Σίνγκ που κινδυνεύει να εκτελεστεί την 31η Μαρτίου, άρα είναι επίγον. Εμείς αγωνιζόμαστε για την κατάργηση θανατικής ποινής και πρέπει κατεπηγόντως να παρέμβει. Σας παρακαλώ να ζητήσετε τουλάχιστον τον κύριο Σούλτς να παρέμβει και να μιλήσει στις ε, Ινδικές Αρχές. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα το φροντίσουμε. Κύριε Κούτας, ζητήστε το λόγο. Α, όχι, ο κύριος ε, Θέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να γραφεί στα πρακτικά εξ ονόματος των 23 ε, Ισπανών βουλευτών της Σοσιαλιστικής Ομάδας ότι θα λάβουμε μέρος ε, στην ψηφοφορία γιατί σε αυτό μας υποχρεώνει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αλλά είμαστε αλληλέγγυοι με τα εκατομμύρια εργαζομένων που απεργούν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Συμμεριζόμαστε τους λόγους της απεργίας ε, διότι τελικά τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα καταπατώνται και ο κοινωνικός διάλογος παραβιάζεται. Είναι δε τα μέτρα τα οποία προτείνονται αντίθετα και με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θέρκας. Κύριε Μπέρμαν, έχετε στήσει και εσείς το λόγο, παρακαλώ. Euh, Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να καταδικάσουμε το πραξικόπημα στο Μαλί. Απερίφραστα να το καταδικάσουμε και να ζητήσουμε αποκατάσταση της αγματικής τάξης στη χώρα αυτή. Επίσης να χαιρετήσω τις δημοκρατικές εκλογές που διενεργήθηκαν στην Σενεγάλη Μάκη Σάλλο, νέο πρόεδρο ε, που εξελέγει, πρέπει να τον συγχαρούμε. Περνάμε λοιπόν τώρα στι ψηφοφορίε. Έκθεση Μορέιρα για το τροποποιημένο καταστατικό στροκανονισμού για το καουτσούκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται έκθεση Taylor